Συγκαρδίνη σχετικά με τη σύναψη της τροποποίησης της Δόχα στο πρωτόκολλο του Κιώτο. Ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Ψηφίσατε, έκλεισε η ψηφοφορία. Μισό λεπτό, μισό λεπτό, το κατάλαβα αυτό που είπατε. Δεν χρειάζεται να υψώνετε τον τόνο της φωνής σας. Εγκρίθηκε η έκθεση. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Κοιτάξτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, παρακαλώ όλους τους βουλευτές να σέβονται τον πρόεδρο και να μην υψώνουν τον τόνο της ε, φωνής τους. Σας το λέω ευθύς εξ αρχής, ε, δεν μου χρειάζονται αυτοί οι οποίοι μιλούν με άσχημο τρόπο, είναι θέμα παιδείας, παιδείας και αγωγής. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι η δεύτερη φορά σήμερα που με αγνοήσατε. Ε, ενώ συμπεριφέρθηκα πολύ καλά, σηκώθηκα και κάλεσα, σας κάλεσα να μου δώσετε το λόγο. Ευγενικά. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στο κεφάλαιο 6 των διαδικαστικών κανόνων. Ε, για τα διαδικαστικά θέματα. Κανόνας 9.1 η αναστολή ή το, ε, η λήξη της συνεδρίας. Ε, σας, ε, ήδη το πρωί σας το ανέφερα και εσείς σηκωθήκατε και φύγατε χωρίς να απαντήσετε στην ερώτησή μου. Αν 40 μέλη της, ε, ε, του Κοινοβουλίου αποφασίσουν να σηκωθούν αυτή τη στιγμή, είμαστε, έχουμε το δικαίωμα να γίνει ψηφοφορία για να λήξει ή να διακοπεί η σημερινή συνεδρία εξαιτία τη διακριτική μεταχείριση που έλαβε χώρα σήμερα εναντίον μα για τη συμφωνία TTIP. Καλό λοιπόν 40 συναδέλφου να σηκωθούν και να ζητήσουν την διακοπή τη συνεδρία. Παρακαλώ 40 άτομα να σηκωθούν αν με υποστηρίζουν. Κοιτάξτε, σήμερα το πρωί το αίτημά σας ή ε, το δικό σας το αίτημα κατατέθηκε όταν είχε ήδη ανασταλεί και διακοπεί η συνεδρίαση. Με βάση το άρθρο 191, όταν 40 βουλευτές, πράγματι μπορούν 40 βουλευτές να ζητήσουν τη διακοπή της συνεδρίασης, εγώ λοιπόν ε, μπορώ να το κάνω αυτό για να διακοπεί η συνεδρίαση και θα το κάνουμε με ονομαστική ψηφορία. Ποιος θέλει να διακοπεί η συνεδρίαση, το ναι σημαίνει διακόπτουμε, το όχι σημαίνει συνεχίζουμε. Ψηφίζετε παρακαλώ, ονομαστική ψηφοφορία, ψηφίζουμε. La Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται η πρότασή σας. Προχωράμε λοιπόν στην ψηφοφορία. Παρακαλώ. Διαδικαστικό. Με βάση το άρθρο 152 και το 190, με την ερμηνεία που δώσατε, το να αποφασιστεί να διακοπεί μια συζήτηση για την επόμενη συνεδρίαση. Αυτό δεν έγινε, δεν ε, ψηφίσαμε επ' αυτού. Γι' αυτό λοιπόν εγώ ζητώ αυτό να αναφερθεί στον κύριο Σούλτς ότι εμείς θέλουμε να γνωρίζουμε διακόπτεται. Δεν υπάρχει διερμηνία ισχυρίζεται η Ευρωβουλευτής και μπορώ να τα πω στα αγγλικά αλλά δεν είναι αλήθεια υπάρχει διερμηνία. Είναι λοιπόν απαραίτητο με βάση τον κανονισμό και ελπίζω τώρα να υπάρχει διερμηνία λέει η βουλευτής. Ελπίζω λοιπόν να ε, τοποθετηθούν όλοι για το πότε θα ψηφίσουμε σχετικά με το TTIP. Αναβλήθηκε η συζήτηση, αλλά για πότε. Δηλαδή θέλω να επενθυμίσω ότι πράγματι είναι το να αναπαιμφθεί στην Επιτροπή ΙΝΤΑ και στην Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να συζητήσουμε και τον Ιούλιο. Και επ' αυτού μπορούμε να ψηφίσουμε. Πρόεδρος, Κοιτάξτε, σήμερα το πρωί δεν ψηφίστηκε το θέμα της αναβολής της συζήτησης. Το μόνο που αποφασίστηκε είναι να αναβληθεί η συζήτηση γιατί η αναβολή της συζήτησης είχε ήδη αποφασιστεί από τον Πρόεδρο. Προχωράμε λοιπόν στην ψηφοφορία. Θα ψηφίσουμε για τη συμμετοχή τη Συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση Ισλανδία όσον αφορά τη συμμετοχή τη Ισλανδία στη δεύτερη περίοδο δέσμευση του πρωτοκόλλου του Κιώτο. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ε, δεν θα σας καθυστερήσω πολύ, για ανθρωπιστικούς λόγους μόνο παρεμβαίνω. Ε, χτες ε, ε, δεν, δεν είδα τον κύριο Σούλτ σήμερα και χτες τον είδα σε κακή υγεία. Μήπως συμβαίνει κάτι μαζί του με την υγεία του, μπορείτε να μας ενημερώσετε. Non mi sembra una... Δεν νομίζω ότι αυτό είναι διαδικαστικό. Ας προχωρήσουμε λοιπόν στην ψηφοφορία με ονομαστική ψηφοφορία για την έκθεση Λαβία παρακαλώ. Ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται το κείμενο. Περνάμε τώρα στην ε, ψηφοφορία τη έκθεση Ζήπελ προσχώρηση τη Κροατία στη Σύμβαση για Μηβαία Δικαστική Συνδρομή Επιποινικών Υποθέσεων. Ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται η έκθεση. Προχωράμε στην έκθεση Χιουσμενόπα, προσχώρηση τη Κροατία στη σύμβαση σχετικά με την καταπολέμηση τη δωροδοκία, στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ονομαστική ψηφορία ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία και εγκρίνεται το κείμενο. Περνάμε τώρα στην έκθεση Λαντσμπεργκης σχετικά με τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας Παράγραφος 1. Το αρχικό κείμενο ψηφίζουμε σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα ποιος είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έλεγχος για το δεύτερο τμήμα. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Αρχικό κείμενο, παράγραφος 2, σε δύο τμήματα για το πρώτο τμήμα. Ε, ονομαστική ψηφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Το, η τρία αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται το κείμενο. Παράγραφος 3, δεύτερο τμήμα, υπέρ παρακαλώ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 11, σε τρία τμήματα, πρώτο τμήμα, υπέρ παρακαλώ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ παρακαλώ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 5, αρχικό κείμενο σε τέσσερα τμήματα. Πρώτο, υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα, Ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται το κείμενο. Τέταρτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 7. Αρχικό κείμενο. Ψηφίζουμε σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα παρακαλώ. Υπέρ, κατά, αποχές Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, ονομαστική ψηφορία, ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται το κείμενο. Παράγραφος 10. Αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 12, αρχικό κείμενο. Σε τέσσερα τμήματα, μια προφορική τροπολογία του κυρίου Μεζέρτσιτς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στην παράγραφο 12 πρέπει να πούμε ανανεώνει την επίκλησή του για την ενίσχυση και παρακολούθηση των ρωσικών δυνατήτων να κάνει προπαγάνδα ειδικότερα στη ρωσική γλώσσα για να εντοπίζει τις κατάλληλες απαντήσεις ε, που θα πρέπει να δίδονται σε μεροληπτικές δηλώσεις σε ευρωπαϊκές γλώσσες. Και έχουμε και τη χρηματοδότηση για συγκεκριμένα project, την παραπληροφόρηση και εδώ συμπεριλαμβάνουμε το εξής, με επαγγελματική αναφορά σε συμφωνία με τη δημοσιογραφική ιδεοντολογία και καλές πρακτικές. Δεν κάνουμε αντίπροπαγάνδα, αντίθετα απαντούμε στη ρωσική ε, προπαγάνδα. Ευχαριστώ. Επιτιμεί κάποιος ε, προφορική τροπολογία από αυτού ή μάλλον ε, υπάρχει κάποιος που να διαφωνεί με αυτή την προφορική τροπολογία. Πάνω από 40 βουλευτές διαφωνούν με την προφορική τροπολογία. Έχετε το λόγο. Γνωρίζοντας ότι το Front National έχει, σχετίζεται με 49 εκατομμύρια που βρίσκονται σε ρωσικές τράπεζες, υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων και πρέπει να τους απαγορευτεί, να, να μην τους επιτραπεί να ψηφίσουν. Η κυρία Λεπέν, νομίζω ότι ε, έχετε ασυλία και την αξιοποιείτε σήμερα για να δυσφημίσετε τους συναδέλφους σας. Είναι σκάνδαλο, είναι σκάνδαλο κύριε. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι το Front National δανείστηκε από ρωσική τραπέζα, ποτέ δεν το έχουμε κρύψει από κανέναν. Όμως, αντιθέτως με εσάς, εμείς δεν εξαγοραζόμαστε μπορεί να είναι μια κατηγορία που σας την επιστρέφω. Βλέπετε τον εαυτό σας στον καθρέφτη όταν λέτε τέτοιες κατηγορίες. Λοιπόν, ψηφίζουμε παρακαλώ. Αρχικό κείμενο για την παράγραφο 12. Το αρχικό κείμενο σε τέσσερα τμήματα ψηφίζουμε. Για το πρώτο τμήμα, ονομαστική ψηφοφορία, ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίθηκε το κείμενο. Το δεύτερο τμήμα με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται το κείμενο. Τρίτο τμήμα, ονομαστική ψηφοφορία Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίθηκε το κείμενο, τέταρτο τμήμα, με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίθηκε το κείμενο. Μετά πάμε στην παράγραφο 12, τροπολογία 12, υπέρ παρακαλώ. Κατά, αποχές, ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ. Ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίθηκε το κείμενο. Παράγραφος 15. Αρχικό κείμενο ε, σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 16. Αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα υπέρ παρακαλώ για το πρώτο. Κατά αποχές εγκρίνεται. Για το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 17. Αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 19, νέο κείμενο, υπάρχει μια προφορική τροπολογία, ε, Έχετε το λόγο. Πρότεινα να προσθέσουμε μια μικρή καινούργια παράγραφο μετά το 19, ως εξής. Υπογραμμίζει για αυτό το θέμα ότι η πρόσφατη τη σαν νομοθεσία για τις ξένες ανευθύμητες οργανώσεις ε, επιτρέπουν στις κυβερνήσεις, στην κυβέρνηση να απαγορεύσει ε, μη επιθυμητές ξένες μη κυβερνητικές οργανώσεις και αυτό είναι ένα ακόμα δείγμα, ανιστικό δείγμα της καταπίεσης ε, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Ευχαριστώ. Είναι πάνω από 40 βουλευτές που διαφωνούν με την προφορική τροπολογία. Περνάμε λοιπόν στην επόμενη προφορική τροπολογία και πάλι της κυρίας Άουταλα, ονομαστική ψηφοφορία. Μισό λεπτό. Πρέπει να την παρουσιάσει. Ναι, πρέπει. Όχι. Έχετε το λόγο. Um, ακόμα πιο ανησυχητικό είναι το γεγονό ότι οι ακροδεξιοί συνάδελφοι μπορεί να αντιτεθούν και ακόμα και με αυτό που θα προτείνω. Προτείνω στην παράγραφο 21 ορισμένες ε, τροποποιήσεις το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί την Κομισιόν να προτείνει νομοθεσία για να εξασφαλιστεί η πλήρη διαφάνεια τη πολιτική χρηματοδότηση και τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τη σύσταση του Συμβουλίου τη Ευρώπη σχετικά ιδιαίτερω με τους, ε, ε, με οικονομικούς και πολιτικούς ενδιαφέροντες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλούμε να ασκηθεί ε, και να εξασφαλιστεί διαφάνεια. Υπάρχει κάποιο που να διαφωνεί παρακαλώ με την τροπολογία. Από ό,τι βλέπω δεν είναι 40 οι βουλευτές που διαφωνούν ως εκ τούτου ψηφίσμα. Ο κύριος Γκόλνης ζήτησε το λόγο. Ήθελα πολύ απλά να ρωτήσω την κυρία Ουτάλα αν με την τροπολογία της ε, στοχεύει επίσης στη χρηματοδότηση των τραπεζών της Αμερικής, της Μέσης Ανατολής, του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και άλλων μερών. Εάν ναι, τότε βεβαίως να τη στηρίξουμε. Uh, Πρόεδρε, ε, σας εγγυώμαι ότι αυτό είναι ένα κάλεσμα για περισσότερη διαφάνεια κάθε ξένης χρηματοδότησης για όλα τα κόμματα. Περνάμε λοιπόν στην ψηφοφορία της προφορικής τροπολογίας με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται το κείμενο. Κατόπιν. Μετά το ε, D, ε, τροπολογία 10, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πάμε στο εκτιμώντας H ε, σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ παρακαλώ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Εκτιμώντας M αρχικό κείμενο υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Εκτιμώντας O αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα αν θέλετε θα κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίθηκε το κείμενο. Θα ψηφίσουμε τώρα για το σύνολο του ψηφίσματος με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίθηκε το κείμενο. Περνάμε στην έκθεση Σαουντάργα σχετικά με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ενεργειακής Ασφάλειας. Μετά την πρώτη παράγραφο, η τροπολογία 5, υπέρ παρακαλώ, κατά αποχές απορρίπτεται. Πάμε στην παράγραφο 7. Αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα ε, ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε ψηφοφορία. Εγκρίθηκε το κείμενο. Παράγραφος 11. Αρχικό κείμενο υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 21. Ε, παράγραφος σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η παράγραφος 24. Αρχικό κείμενο σε τέσσερα τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι απορρίφθηκε ηλεκτρονική επαλήθευση για το δεύτερο τμήμα του 24 ψηφίζουμε παρακαλώ έκλεισε ψηφοφορία απορρίφθηκε το κείμενο τρίτο τμήμα υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. Τέταρτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Επαλήθευση για το τέταρτο τμήμα. Εντάξει. Ε, ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Παρακαλώ να σκόντε τα χέρια σας, γιατί δεν βλέπω κι εγώ καλά. Πάμε στην παράγραφο 25, σε δύο τμήματα, πρώτο τμήμα, υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονική επαλήθευση, ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία εγκρίθηκε με νέα ψήφους διαφορά. Παράγραφος 32, αρχικό κείμενο, ονομαστική ψηφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίθηκε το κείμενο. Έβαλα και τα γυλιά μου να βλέπω καλύτερα, αλλά δεν φταίω εγώ γιατί δεν καλά τα χέρια. Πάμε στο επόμενο. 32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 33. Η παράγραφος 33 κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλειση ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Η 34. Αρχικό κείμενο, ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται το κείμενο. Επειδή λοιπόν εδώ στην ψηφοφορία είναι μικρές οι διαφορές, σας παρακαλώ πολύ να σηκώνετε καλά τα χέρια γιατί μετά είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε ηλεκτρονικές επαληθεύσεις. Πρέπει να είναι 38 αρχικό κείμενο υπέρ, για το πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές, το δεύτερο τμήμα, μισό λεπτό, εγκρίνεται, εγκρίνεται. Εντάξει λέει ο Πρόεδρος. Δεύτερο τμήμα τώρα, υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι απορρίφθηκε ηλεκτρονική επαλήθευση για το δεύτερο τμήμα της 38. Έκλειση Έκλεισε ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Μετά την 38, τροπολογία 6, ε, ψηφίζουμε με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίφθηκε το κείμενο. Μετά την παράγραφο 39, τροπολογία 1, σε, δύο, σε με ονομαστική ψηφοφορία ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Το κείμενο εγκρίθηκε. Η 40 ε, αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα για το πρώτο υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται για το δεύτερο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 41 αρχικό κείμενο πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές Νομίζω ότι απορρίφθηκε ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίζουμε για το δεύτερο τμήμα τη 41. Έκλειση ψηφοφορία. Εγκρίθηκε το κείμενο. 43. Αρχικό κείμενο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 44 αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα. Θέλετε ηλεκτρονική επαλήθευση για το αρχικό κείμενο του 43. Εντάξει, επαλήθευση για τη 43, για το αρχικό κείμενο. Ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίθηκε το κείμενο. Πάμε τώρα στη 44, αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές Νομίζω ότι εγκρίθηκε η ηλεκτρονική επαλήθευση για το δεύτερο τμήμα τη 44 ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται ή εγκρίθηκε. Μετά τη 44 η 2 ονομαστική ψηφοφορία ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίφθηκε το κείμενο. Η 45 αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Ονομαστική ψηφοφορία, Ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίθηκε το κείμενο. Δεύτερο τμήμα. Ονομαστική ψηφοφορία, Ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίθηκε το κείμενο. Παράγραφος 49 υπέρ κατά αποχές 49 σε δύο τμήματα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Για το δεύτερο τμήμα τη 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 55 αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 58 αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ηλεκτρονική επαλήθευση γιατί ξέρετε υπάρχουν πάρα πολλοί βουλευτές που δεν σηκώνουν καλά το χέρι τους και είναι δύσκολο για μένα γιατί η διαφορά είναι μεταξύ 10 και 15 ψήφων. Σας παρακαλώ πολύ να σηκώνετε καλά το χέρι σας. Έκλεισε τώρα η ψηφοφορία. Εγκρίθηκε το κείμενο. Η παράγραφος 60, αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα, πρώτο υπέρ, κατά, αποχές, απο... εγκρίνεται, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται ή 61. Λοιπόν, ηλεκτρονική επαλήθευση για το δεύτερο τμήμα της 60. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Η 61. Αρχικό κείμενο. Ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίθηκε το κείμενο. Η 68 αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 71 αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 73 αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 74 αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 77 αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, ονομαστική ψηφορία, ψηφίζουμε για το δεύτερο τμήμα της 77. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίθηκε το κείμενο. Η 78 αρχικό κείμενο ονομαστική ψηφοφορία ψηφίζουμε. Εγκρίνεται το κείμενο. Η 79 για το πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η 80 αρχικό κείμενο υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η 83 αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα υπέρ για το πρώτο, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Η 84 αρχικό κείμενο ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 87 αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίθηκε το κείμενο. 90. Αρχικό κείμενο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 91. Αρχικό κείμενο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 92. Αρχικό κείμενο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 94. Αρχικό κείμενο. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 102 αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 103 αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 110 αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται μετά την 111 την παράγραφο η τρία ψηφίζουμε μονοστική ψηφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφορία. Απορρίφθηκε. Η επτά, Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Μετά τη 116 αρχικό κείμενο, πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 117 αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 118 αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα πρωτοτμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίθηκε το κείμενο. Παράγραψε 119. Αρχικό κείμενο υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 124. Αρχικό κείμενο. Ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίθηκε το κείμενο. Η 125 αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 127 αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 129 αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 130 αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 131 αρχικό κείμενο ονομαστική ψηφορία ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίθηκε το κείμενο. Η 132 αρχικό κείμενο υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 133 αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 139 υπό, υπότιτλος, η επικεφαλίδα μάλλον, αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την 141 αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα τώρα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, η 143 αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 145 αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 151 αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 152 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 155 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 156 Αρχικό κείμενο υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ε, εκτιμώντας β, αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Εκτιμώντας H, αρχικό κείμενο υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται εκτιμώντας ή αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Εκτιμώντας J, αρχικό κείμενο ε, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Εκτιμώντας K, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Εκτιμώντας Ερ. η τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ. Ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία απορρίφθηκε το κείμενο. Εκτιμώντας τι αρχικό κείμενο υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία εγκρίθηκε, είχατε δίκιο εσείς. Εκτιμώντας γιου, αρχικό κείμενο, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Εκτιμώντας ύψιλον, αρχικό κείμενο υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Κονσιντεράντο Z, αρχικό κείμενο, μονομαστική ψηφοφορία, ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Το κείμενο εγκρίθηκε. Εκτιμώντας AB, αρχικό κείμενο υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Εκτιμώντας AC, ε, αρχικό κείμενο υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Εκτιμώντας AD, ε, αρχικό κείμενο υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Εγκρίνεται, λέει ο πρόεδρο. Εντάξει, αν θέλετε να τα λέω πιο αργά. Λοιπόν, εκτιμώντας ή e σε δύο τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Εκτιμώντας AG αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται εκτιμώντας AK αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται εκτιμώντας AQ ο κύριος Γκόλνης έχει το λόγο παρακαλώ Κύριε Πρόεδρε για το άρθρο 75 του κανονισμού. Αυτό θέλω να επικαλυστώ, το οποίο επιτρέπει στον πρόεδρο της συνέλευσης να παραπέμψει ένα κείμενο στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή όταν υποβάλλονται πάνω από 50 τροπολογίες κατά τμήματα είναι η περίπτωσή μας αυτή. Και ο Πρόεδρος δεν, αυτό το, δεν άσκησε αυτό το προνόμιο που έχει. Αναρωτιέμαι λοιπόν, και το αναρωτιούνται πολλοί συνάδελφοι, το ίδιο προνόμιο άσκησε για την έκθεση που έπρεπε να εξετάσουμε σήμερα το πρωί. Ε, είναι ύποπτο λοιπόν ε, το ότι δεν ασκεί το ίδιο προνόμιο για αυτή τη συγκεκριμένη έκθεση και αυτό το καταθέτω προς προβληματισμό όλων. Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ αργά για να θίξετε αυτό το θέμα. Με πάση περιπτώσει, το θέμα είναι όπως είπατε στην διακριτική ευχαίρεια του Πρόεδρου. Ε, εγώ, ο Πρόεδρος, αποφασίζω ότι ψηφίζουμε. Λοιπόν, ψηφίζουμε για το αρχικό κείμενο AQ υπέρ παρακαλώ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και τώρα θα ψηφίσουμε για το σύνολο του ψηφίσματος με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίφθηκε το κείμενο, το ψήφισμα. Ich wollte η κυρία Μάγερ, θα ήθελα να ενημερώσω λίγα του αδέλφου που είναι οι παρακαθήμενοι μου, γιατί αν είχαν προσέξει στην ψηφοφορία, ήταν πολύ λίγε ε, οι τροπολογίε και κυρίω για το αρχικό κείμενο. Δεν ήταν ουσιαστικέ τροπολογίε. Λοιπόν, άλλη φορά να κοιτάτε λίγο καλύτερα τον κατάλογο ψηφοφορία που σα έχουν καταθέσει. Πρόεδρος, πάμε στην ετήσια έκθεση της Επιτροπής Εποπτείας της Όλαφ για το 2014 και ψηφίζουμε για την πρόταση, κοινή πρόταση ψηφίσματος που έχει κατατεθεί από τρεις πολιτικές ομάδες. Ψηφίζουμε λοιπόν με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Η ψηφοφορία έκλεισε εγκρίθηκε το κείμενο. Το ψήφισμα εννοεί ο πρόεδρος. Πάμε τώρα στην κατάσταση στην Ουγγαρία. Προτάσεις ψηφίσματος από τέσσερις ομάδες. Σε παράγραφος 3 αρχικό κείμενο ψηφίσμα σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίζουμε. Έκλεισε ψηφοφορία. Εγκρίθηκε το κείμενο. Σας παρακαλώ πολύ εσείς που είστε από εδώ από αριστερά να σηκώνετε το χέρι σας κανονικά γιατί δεν μπορώ να βλέπω, δεν σας βλέπω καλά, δεν ξέρω τι ψηφίζετε. Δεύτερο τμήμα τώρα ψηφίζουμε υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η παράγραφος 5, αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα, υπέρ παρακαλώ για το πρώτο τμήμα, υπέρ, υπέρ για το πρώτο τμήμα, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 9, αρχικό κείμενο, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 10. Όχι, ηλεκτρονική επαλήθευση για την ενέα αρχικό κείμενο ψηφίζουμε παρακαλώ. Εγκρίθηκε το κείμενο. Παράγραφος 10. Αρχικό κείμενο υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 11. Αρχικό κείμενο σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ παρακαλώ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τώρα, ηλεκτρονική επαλήθευση για το δεύτερο τμήμα της 11. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίθηκε το κείμενο. Το τρίτο τμήμα της 11 υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 12. Αρχικό κείμενο ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. Στο F, λατινικό, ποιοι είναι υπέρ. Για την παράγραφο 12 θα υπάρξει ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραστη στις Δεκτό το κείμενο. Γυρνάμε στο F λατινικό. Πρώτο τμήμα. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Δεύτερο τμήμα. Ποιοι είναι υπέρ Κατά. Αποχές. Δεκτό. Το σύνολο του ψηφίσματος, τροπολογημένο, έχει ζητηθεί ονομαστική ψηφοφορία η οποία αποσύρθηκε. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Πρέπει να σηκώνετε τα χέρια σας γιατί αλλιώς θα υπάρξει ηλεκτρονικός έλεγχος. Λοιπόν, ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Καλά ακούω. Πέρα στις ψηφοφορίες. Το κείμενο γίνεται δεκτό. Ψάχνω το επόμενο. Πρόταση ψηφίσματο μετά την παράγραφο 3 έχω την τροπολογία 31 για την Τουρκία. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχέ, δεκτή. Στην 9, την 24, ονομαστική ψηφοφορία ψηφίζουμε. Πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Μετά την παράγραφο 15 έχω την 28. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 37. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 30 μετά την 16. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 15. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ονομαστική ψηφοφορία. Υπέρ. Πέραση της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 32. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 33 στην 29 ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Μετά την 30 έχω την 9 ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 17 ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 4 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Ένα. Έχει καταπέσει ένα. 34 στην παράγραφο 33. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 18 υπέρ. Έχει καταπέσει και αυτή. 38. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Ηλεκτρονικός έλεγχος λοιπόν για την 38. Βοτοκιούσα. Τέλος της ψηφοφορίας. Απερίφθη. Πέντε υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Στην 35, την παράγραφο 3... Α, α, όχι, όχι, γυρνάμε στην 5 έλεγχος για την 5. Πέρα στις ψηφοφορίες δεκτό το κείμενο. Κοιτάξτε, έχω φορές τα γυαλιά μου, βλέπω. Λοιπόν, στην παράγραφο 35 έχω την τροπολογία 35 Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση η ψηφοφορίας. Το κείμενο γίνεται δεκτό. Στην 36. Έχω τη 19. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Στην 37 έχω την 20. είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 36 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Στην 38 το αρχικό κείμενο σε τρία τμήματα. Το πρώτο, σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Στην 39 την 26 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Στην παράγραφο 42 την 21 ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 44 την 22 ονομαστική ψηφοφορία ψηφίζεται. Λοιπόν, πρώτο τμήμα τη 44 ψηφίζουμε. Κατά. Αποχέ. δεκτό. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχέ. δεκτό. Μετά τη 44 έχω την τροπολογία 7. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχέ. Νομίζω ότι έγινε δεκτή, αλλά θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την 7. Λοιπόν, δεκτό. 23. Ονομαστική ψηφοφορία ψηφίζεται. Πέρασε ψηφοφορίες, Δεκτό. Έχω την 27 τώρα, ονομαστική ψηφοφορία και για την 27 ψηφίζεται. Πάτε αργά, έχετε κουραστεί, τεμπελιάζετε. Πέραση ψηφοφορία. ψηφοφορίας. Απερίφθη. Τροπολογία 2, ονομαστική ψηφοφορία ψηφίζεται. Απερίφθη. 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Αν δεν σηκώνετε τα χέρια δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, ηλεκτρονικός έλεγχος για την 12 ψηφίζεται. πέρα στις ψηφοφορίες. Δεκτό. 13. Και είναι υπέρ της 13. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Στο Β έχω την προφορική τροπολογία Σόμερ. Υπάρχει μια προφορική τροπολογία η κυρία Ζόμερ. Λειτουργεί το μικρόφωνο σας, μάλιστα, τώρα είναι εντάξει. Ε, η τεχνολογία. Ε, πρόεδρε, προτείνω να διορθώσουμε ένα σφάλμα στην επόμενη πενταετία να το αντικαταστήσουμε με τους όρους στην παρούσα θητεία. Το έχω συμφωνήσει με την εισηγήτρια και παρακαλώ να το υπερψηφίσουμε. Να μην μιλάμε για πενταετία αλλά για τη θητεία αυτή. Και a favore Ποιοι είναι υπέρ της προφορικής. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Στο ΚΑΠΑ έχω την 14. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Μετά το ΚΑΠΑ έχω την 29 ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. πέρα της ψηφοφορίας. Δεκτό. Τώρα το ψήφισμα στο σύνολό του, ονομαστική ψηφοφορία ψηφίζεται παρακαλώ. Il voto è chiuso. Πέρα στις ψηφοφορία γίνεται δεκτό το κείμενο. Θα περάσουμε τώρα στις